αίτηση άρση τη κοινοβουλευτική ασυλία τη κυρία Ίγκεμπορ Γκρέσλε στα πλαίσια κριτική διαδικασία σε βάρο τη. Οι αρμόδιε γαλλικέ αρχέ μου απίφθηναν αίτηση άρση τη κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Στίβα Μπριούα στα πλαίσια προκαταρκτική έρευνα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι εν λόγω αιτήσει παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου. Έλαβα από